με τις προσπάθειές μας ε, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση ως προς την προστασία των ε, θεμελιωδών ελευθεριών και των προσωπικών δικαιωμάτων στο Θιβέτ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγη εδώ η συζήτηση για αυτό το θέμα. Αξιότιμοι συνάδελφοι, επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι παρεμβάσεις του ενός λεπτού σύμφωνα με το άρθρο 150. Το άρθρο 150 προβλέπει πώς μπορούμε να αφιερώσουμε το πολύ 30 λεπτά σε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε άνω των 74 ετοιμάτων. για να λάβουν οι συνάλφοι τον λόγο. Οπότε είναι προφανές 74 μονόλεπτα επί 30 λεπτά δεν βγαίνουν. Οπότε υπήρξε μια επιλογή των όσων θα μιλήσουν με σαφή κριτήρια, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήδη σε άλλη συζήτηση ε, δεν έλαβαν την προηγούμενη φορά τον λόγο για ένα λεπτό θα μιλήσουν τώρα ενώ αυτοί οι οποίοι στο παρελθόν είχαν ήδη μιλήσει σε προηγούμενη συζήτηση δεν θα λάβουν τον λόγο και όσοι δεν είχαν λάβει και δεν θα λάβουν τον λόγο ε, ειδοποιήθηκαν με email για να μην έρθουν άσκοπα και περιμένουν να μιλήσουν. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε έτσι να έχουμε μια λογική συζήτηση. Οπότε, όπως σας είπα, αυτή είναι η διαδικασία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα μιλήσει ο κύριος Σβένσον. Ευχαριστώ. Στις 11 Απριλίου ε, υπήρχαν ε, συναντήσεις ανάμεσα στο Κοινοβουλίο και το Σουδάν και ήταν οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές και παρακολουθήσαμε ε, με, ιδιαίτερη, ε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εκλογές. Ο πρόεδρος, ο κύριος Μπασίρε, κατηγορήθηκε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλοι γνωρίζουν την καταστολή που έχει βάλει στο Σουδάν και μόνο το περασμένο μήνα στο Νότιο Σουδάν ε, σκοτώθηκαν 400 άνθρωποι ε, και ε, Επίσης απείλησε ο κύριος Μπασίρε να εκδιώξει από το Σουδάν τους όσους συμμετέχουν στις διεθνείς ερευνευτικές δυνάμεις και θα πρέπει να Γνωρίζουμε επίσης ε, ότι έχουν δοθεί 1,4 εκατομμύρια στο Σουδάν ε, για, ε, ως βοήθεια νοικοδόμησης. Σας ευχαριστώ. Εδώ πέρα τελείωσε ο χρόνος σας. Κύριος Μπαλτσίτης. Oh, Μπαλτσίτης. ναι. Κύριε Μικολέγκος, Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούμε τώρα φωνές που λένε πως ανακάμπτει η ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά δεν έχει τελειώσει η κρίση. Σε πολλά κράτη-μέλη μιλάμε μόνο για τα δημόσια οικονομικά, όμως η ανεργία αυξάνεται και έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα. Περιέργως, ε, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενούν κράτη-μέλη για επιτυχίες, ενώ αυξάνεται η ανεργία. Η κοινωνική κάλυψη μειώνεται και οι άνθρωποι που, που είναι φτωχοί αυξάνονται. Οι άνθρωποι αυτοί δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταπολέμηση ή αύξηση της φτώχειας. Δεν νομίζω ότι αξίζει να επενούμε και κυβερνήσεις όταν αυξάνεται η ανεργία, πρέπει να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βγούμε από την κρίση και να δούμε τι κάνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις στους ανθρώπους. Κυρία Αλφάνο. Σας ευχαριστώ. 16 άτομα έχουν καταδικαστεί στο ε, Ιταλικό Κοινοβούλιο και δεν υπάρχει νόμος ε, βεβαίως ε, που να απαγορεύει σε κάποιον που έχει καταδικαστεί από τον εκλεγή βουλευτής. Τώρα λοιπόν στην Ιταλία έχουμε αυτό το λεγόμενο καθαρό κοινοβούλιο θα πρέπει νομίζω, τουλάχιστον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να είναι κάποιο υποψηφίο, να μην έχει ποινικό μητρό. Στο παρελθόν είχαμε δε εξετάσει την περίπτωση Καζίνη και τελικά είπαμε πως η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων δεν θα μας ασχολήσει αυτό το θέμα αλλά το άρθρο 119, το 123 σημαίνει πως θα πρέπει να δούμε να έχουμε κοινά, κοινούς κανόνες για να εκλεγεί κάποιος. Η κυρία Γκρέζ. Ε, καλησπέρα. Το αεροδρόμιο Φόνταραμπή θεωρείται ως το πλέον επικίνδυνο της χώρας από την πολιτική αεροπορία γιατί η διάδρομη απογείωσης και προσγείωσης είναι πάνω από Διάντε ε, Ντερούν. κοντά στα ισπανικά σύνορα επίσης δεν τηρείται η νομοθεσία για το χρόνο απογείωσης. Ε, είναι επικίνδυνο για όσους μένουν στις μεθόριες περιοχές και ε, θέλουμε να ξέρουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζει την καταστροφή δηλαδή φυσικών βιοτόπων που προστατεύονται βάσει της ε, σχετικής οδηγίας μα έχει η ίδια χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση αυτών των περιοχών ε, και στο Σαν Σεμπαστιά στη χώρα των Βάσκων υπάρχει ήδη αεροδρόμιο δεν χρειάζεται να θέτουμε σε κίνδυνο τέτοιες ευαίσθητες περιοχές και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα μεταφορές για να υπάρξει διασύνδεση με το BRI e. Πότε θα αποφασιστεί λοιπόν η επέκταση των υπάρχοντων δικτύων. Ευχαριστούμε ο κύριος Μιγκάλης και τώρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την ε, δολοφονία του Μάξιμ Ντουγιέφ, Ρώσου δημοσιογράφου στο Καλίνιγκραντ. Ε, ήταν ένας μπλόγκερ, γνωστός δημοσιογράφος και δεν είναι η πρώτη περίπτωση δολοφονίας δημοσιογράφου στη Ρωσία από το 2002. Τουλάχιστον 10 τέτοιες πολιτικές δολοφονίες μειώθηκαν. Είναι ανησυχητικό το φαινόμενο. Ε, δεν υπάρχει ελευθερία για τους δημοσιογράφους, δεν μπορούν να εργαστούν. Ε, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό στον ευρωσικό διάλογο. Θα κάνουμε σεμινάριο ε, στο Κοινοβούλιο αν υπάρξει συμφωνία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Πρέπει να συζητήσουμε με τους ομολόγους μας και να τονίσουμε ότι η προστασία της ελευθερίας έκφρασης των δημοσιογράφων πρέπει να αποτελέσει αίρισμα του πολιτικού διαλόγου μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Κουντής. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας αναφέρω το γεγονός ότι πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι Αμερικάνοι εισαγγελείς κατήγγυλαν κατηγορίες εναντίον της γερμανικής εταιρείας Daimler για δωροδοκία ξένων αξιωματούχων προκειμένου να εισπράξει και να υπογράψει κρατικά συμβόλαια. Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι η επιχείρηση είναι αναμεμειγμένη σε μακρόχρονη διαδικασία δωροδοκιών το ίδιο θέμα είχε προκύψει και με τη siemens η οποία ακολούθησε την ίδια πρακτική και διήφθηρε τις κυβερνήσει 30 χωρών προκειμένου να έχει προμήθειε στι δημόσιε επιχειρήσει. Ένα σκάνδαλο που εξακολουθεί να συγκλονίζει και την Ελλάδα. Κατόπιν τούτου, εκτό από τη χρηματοπιστωτική κρίση, έχουμε και κρίση ηθική. Η γερμανική κυβέρνηση μέχρι πρόσφατα δεν καταδίωκε τη δωροδοκία εκτό των συνόρων, επροσποιείται ότι δεν ήξερε τα γεγονότα. Τέλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντί να ενεργήσει αντί να ενεργοποιήσει την ε, επιτροπή κατά της απάτης δεν υπερασπίζεται την νομιμότητα και σε πολλές περιπτώσεις δεν περιφρουρεί τα χρήματα των ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Σαλαβράκος. Κυρία Πρόεδρε, οφείλω να καταγγείλω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι σήμερα στις 2 και 4 το πρωί η τουρκική κορβέτα Μπάφρα παρεβίασε 18 μίλια μόλις από τις ακτές της Αθήνας τα ελληνικά χωρικά ύδατα και μάλιστα εζήτησε να κάνει νιοψία σε παραπλέον ελληνικό εμπορικό πλοίο. αποδεικνύεται λοιπόν ότι όσα λέχθησαν στο πρώτο μέρος της συζητήσεως σχετικά με το λεγόμενο οικονομικό πρόβλημα της ελλάδος είναι όχι τόσο ακριβή. κυρίως το, πρόβλημα της ελλάδος είναι πολιτικό. προέρχεται από το γεγονός ότι η γειτονική αυτή χώρα απειλεί κάζους μπέλικα της ελλάδος και προκαλεί συστηματικά ε, τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις όχι μόνο με παραβιάσεις των ε, υδάτων αλλά και του εναέριου χώρου. Το μικρόφωνο έχει σβήσει του κυρίου Σαλαβράκου. Entschuldigung, da ist ein Mikro. Με συγχωρείτε, είχε σβήσει το μικρόφωνο σας. Παρακαλώ. Πρέπει να γίνει γνωστό ότι η Ελλάδα έλαβε αυστηρά μέτρα που σε τελευταία ανάλυση καταπνίγουν στην κυριολεξία τα ελληνικά νοικοκυριά και οι Έλληνες πλέον είναι εκτός των ορίων τους. Έχει εξαντλήσει τις αντοχές της ελληνικής κοινωνίας και τις οικονομικές αντοχές των Ελλήνων. Το πρόβλημά της, όπως είπα, είναι κυρίως πολιτικό. δεν ζητάμε χρήματα από κανέναν ευρωπαίο πολίτη. ζητούμε τη συμπαράσταση της ευρωπαϊκής ένωσης σαν οντότητας τρόπον ώστε να ξεπεράσουμε τις αριθμίες αυτές των αγορών που επιτίθενται κατά του ευρώ. Σας ευχαριστώ. Παρά το τεχνικό πρόβλημα εξαντλήθηκε ο χρόνος σας. Ο κύριος κατόπιν. πριν από δέκα χρόνια επέβαλαν ε, τότε οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρώσεις κατά της ε, χώρας μου της Αυστρίας η οποία δεν μπορούσε να συμμετάσχει στα συμβόλαια στα συμβούλια με αλλά ε, αναγκαζόταν μόνο να πληρώνει και δεν ε, παρουσίαζε νομίζω κανένα κίνδυνο για την ε, δημοκρατία. Αντιθέτως ε, επρόκειτο για επέμβαση στην κυριαρχία της Αυστρίας. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να σεβόμαστε την κρατική κυριαρχία των κρατών μελών και την πολιτική άποψη των λοιπόν. Και ελπίζω πως ο κύριος Λουί Μισελ ο οποίο είχε ξεκινήσει τότε αυτή την πρωτοβουλία, να μπορεί τώρα να κάνει ελεύθερος διακοπές στην Αυστρία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ματιέ κατόπιν έχει τον λόγο. Πρόεδρε, εχθές ε, η Γαλλία απέτησε φόρο τιμή ε, σε έναν αστυνομικό, τον κύριο Νεγά, επικεφαλής ε, μονάδας που δολοφονήθηκε από την ΕΤΑ στι 16 Μαρτίου σε ανταλλαγή πυρών στο Παρίσι. Ευθύνεται η ΕΤΑ εδώ και 40 χρόνια για το θέμα των 830 ατόμων και πρώτη φορά όμως επιτίθεται σε Γάλλο αστυνομικό. Με αυτή τη δολοφονία πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οφείλουμε να καταπολεμήσουμε την ε, τρομοκρατία. Η γαλλοϊσπανική συνεργασία σε αυτό το τομέα θα αποτελέσει υπόδειγμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ελπίζουμε. Η Γαλλία ήταν ένα από τα πρώτα κράτη-μέλη που συγκρότησε κοινέ δυνάμει στο ε, κοινό ευρωπαϊκό χώρο ασφάλεια, ε, ζήτησε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη και απεδείχθη αποτελεσματική η δράση τη. Δυστυχώ όμω δεν μπόρεσαν δεν μπόρεσε αυτή η αστυνομική και δικαστική συνεργασία να αποτρέψει τη δολοφονία δολοφονία πρέπει να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία για να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικότερα την τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζο Χίγκιν. Κυρία Πρόεδρε, εγώ ή ο κύριος, εσείς, εσείς κύριε Χίγκινς, εσείς ε, αργότερα. Τζο, Τζο Και να με συγχωρείτε, λέει η πρόεδρος. Εάν μπορείτε να μηδενίσετε το χρόνο. Ο πρόεδρος της κίνησης ε, των πολιτών την, ε, Σουζ, της ε, κοιλάδας Σούζα προσπαθεί να σταματήσει την οικοδόμηση μια γραμμής ε, σιδηροδρομικής υψηλή ταχύτητας. Σε μια πολύ στενή κοιλάδα με βάθος μόνο 21 χιλιόμετρα υπάρχει ήδη και αυτοκινητόδρομος και άλλη μια σιδηροδρομική γραμμή. 48% μόνο της ε, δυναμικότητα του σιδηρόδρομου χρησιμοποιείται. Εν τω μεταξύ τι θα γίνει, θα μολυνθεί η περιοχή και από αμίαντο και από ουράνιο κατά τη διάρκεια των εξκαφών. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν κινητοποιηθεί. Χρησιμοποιείται αστυνομική βία για να σταματήσει αυτή η εκστρατεία. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει τη χρηματοδότηση του έργου και να ακυρωθεί το έργο. Οι άνθρωποι εκεί δεν θα φοβηθούν και διώκονται γιατί είναι υπέρ της κοινής λογικής και του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ. Νάταλ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ανησυχώ όλο ένα και περισσότερο για τον τρόπο που τα τομικά συμβούλια στην βορειοδυτική Αγγλία χρησιμοποιούν τα τέλη από τα αυτοκίνητα για να αυξήσουν τα εισοδήματά τους. Στην πόλη παραδείγματο χάρη ε, είναι σχεδόν χωριό και τι χρεώνουν τη στάθμευση των αυτοκινήτων ε, και ε, για να αυξήσουν το εισόδημά τους ε, και το αποτέλεσμα είναι να χρεοκοπούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλοι δείχνουμε το δάχτυλο το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά συγγνώμη θα πρέπει να δούμε γιατί έχει προβλέψει σχετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχουμε ένα νομικό πλαίσιο στην οδική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010. Να η ευφυΐα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικά όλοι δακτυλοδειχτούν άλλους υπευθύνου αντί να απορρίπτουν τις ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η πραγματική υπέτεια. Ευχαριστούμε κυρία Σινκλέρ. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ προέρχομαι από τα Green... από τα West Midlands και έχουμε προσπαθήσει να προστατεύσουμε αυτή την πράσινη ζώνη από τον οικισμό. Όμως η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αρχίσει να οικοδομεί κατοικίες εκεί πέρα. Υπάρχει έλλειψη σεβασμού των παραδόσεων. Αλλά τι σας νοιάζει εσάς από όταν μπήκε το Ηνωμένο Βασίλειο μας αγνοείται εμάς και τις παραδόσεις μας και τίποτα άλλο δεν περιμένω από εσάς. Ο κύριος Αντωνέσκου τώρα. Η κυρία Αντωνέσκου. Ευχαριστώ θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρωμένη πολιτική για την καταπολέμηση της ε, βίας ε, που υφίστανται οι γυναίκες. Ε, έχει συζητηθεί ε, αυτό το θέμα εν πολλής, αλλά δεν υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στις ε, πολιτικές ομάδες. Ε, και το θέμα όμως της οικογενειακής βίας δεν μπορεί να γίνει πολιτικό θέμα. Πρέπει να επικρατήσει η δικαιοσύνη στην κοινωνία μας και μην ξεχνάτε ότι πέρα από την σωματική υπάρχει και η ψυχολογική βία κατά των γυναικών. Ε, χαιρετίζω το ότι η Ισπανική Προεδρία έχει αναδείξει σε προτεραιότητα το θέμα της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, αλλά πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες. Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την καταπολέμηση της βίας, ε, η τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας είναι θετικά βήματα. Ευχαριστώ, η κυρία ούτε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασχοληθεί με τη φτώχεια και είπε πως φέτος είναι το Ευρωπαϊκό Ότος Καταπολέμησης Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Έχουμε πολλά εκατομμύρια Ευρωπαίους που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας άνθρωποι που έχουν και δουλειά δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει για συγκεκριμένες δράσεις το 2010 17 εκατομμύρια ευρώ για σεμινάρια, δημόσιες διαβουλεύσεις ε, για να καταπολεμήσουν τα στερεότυπα. Καλή αυτή η πρωτοβουλία αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθούν με διάφανο τρόπο αυτά τα κονδύλια για να πάνε στους πραγματικά απελπισμένους. Δεν φτάνει επίσης αυτό για την καταπολέμηση της στόχιας. Πρέπει η Ένωση και τα κράτη-μέλη να λάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις για να υπάρχει σωστή κατανομή των κονδυλίων σε αυτούς που τα χρειάζονται. Ευχαριστώ κύριε Στούσας. Η της Ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει το σχέδιο για την κατασκευή 1.600 νέων κατοικιών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ την επέκταση του επικισμού στη δυτική όχθη τη συνέχιση του αποκλεισμού της λωρίδας της γάζας και γενικότερα την κλιμάκωση των επιθέσεων του ισραηλινού στρατού στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, αποκαλύφθηκε στον πιο δύσπιστο τα εγκληματικά σχέδια του ισραήλ και γενικότερα των υπεριαλιστών ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στους λαούς της ευρύτερης περιοχής. το ισραήλ εξαπολύει νέο γύρο δολοφονικών επιθέσεων σε βάρος του παλαιστινιακού λαού έχοντα εξασφαλίσει τη στήριξη και αναβάθμιση των σχέσεών του με την ευρωπαϊκή ένωση της ηπα και το νατο σε συνθήκες έντασης των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών στο κουαρτέτο. στήριξη που με ιδιαίτερη έμφαση και ζήλο επανέλαβαν οι ηνωμένε πολιτείε τη αμερική κατά τη διάρκεια τη πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού του ισραήλ σε αυτή τη χώρα τονίζοντα ότι το ισραήλ είναι κάτι παραπάνω από πρώτη προτεραιότητα για τα γεωστρατηγικά υπεριαλιστικά σχέδια των ηπα στην ευρύτερη περιοχή. Παλεύουμε με για τη δημιουργία. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο χρόνο σα τελείωσε. Ο κύριο Πάσκα κατόπιν είναι ο επόμενο ομιλητή. Κύριε Πάσκα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Στην Ουγγαρία υπάρχουν γύρω στους 400.000 Σλοβάκους όπως ακριβώ υπάρχουν και 400.000 Ούγγροι στην Σλοβακία. Η Ουγγρική μειονότητα στην ε, Σλοβακία, όπως σας είπα, είναι σε μεγάλο αριθμό, παρόλα αυτά έχει, ήταν, αλλά έχει μειωθεί σε ένα δέκατο του αρχικού μεγέθους της, γιατί δεν υπάρχει εκπαίδευση στην ε, μητρική τους γλώσσα εξού και Βεβαίως οι πρόσφατες ε, επικρίσεις από τον πρόεδρο της Ουγγρικής Μειονότητας καθώς υπάρχει καταπίεση της ε, μειονότητας κατά το οποίο είναι κοινικό Σλοβάκοι, Σέρβοι και Ρουμάνοι ενδιαφέρονται για τις, ε, για τις μειονότητες ο δε εκπρόσωπος πολίτη λέει πω στην Ουγγαρία υπάρχει πλήρη αφομοίωση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ Νικολέσκου κατόπιν. Κυρία Πρόεδρε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αυστηρά μέτρα για την τροφιμική ασφάλεια και οι παραγωγοί πρέπει να κάνουν ένα σωρό προσπάθειες για να σέβονται αυτούς τους κανόνες αλλά πάνω από 75% των κοτόπουλων και των και των κοτών που καταναλώνονται στην Ευρώπη είναι μολυσμένα. Τρία στα τέσσερα κοτόπουλα των ευρωπαϊκών πτυνοτροφίων υποφέρουν από σαλμονέλα. Ρωτώ λοιπόν, τι να κάνουμε ούτω ώστε οι Ευρωπαίοι να, να τρώνε υγιή τρόφιμα και τρόφιμα ποιότητας και αυτοί οι σκληροί κανόνες που έχουμε είναι πραγματικά οι καλύτεροι. Ο κύριος Σταμπάτζη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα η ΚΟΑ κρασιού του 2007 ενημερώνεται στις διάφορες χώρες αλλά έγινε μία παραβίωση των διατάξεων διότι η Κομισιόν και κατόπιν ετήματος της Σλοβακίας κατέταξε το τοκάι ως κρασί προέλευσης ντόπ και, ως ε, και ταυτόχρονα γεωγραφικής προέλευσης. Ή στη μία κατηγορία θα ανήκει αυτό το κρασί ή στην άλλη. Δεν γίνονται και τα δύο είναι παράνομα. Το σλοβακικό αίτημα δεν αφορά την, γεωγραφική, την εγκυμένη γεωγραφική προέλευση. Υπάρχει ένας νόμος όμως στη Σλοβακία για το κρασί που δεν εφαρμόζεται. Και ρωτώ την Κομισιόν, ζητώ μάλλον από την Κομισιόν, να σταματήσει αυτή την κατάσταση παραβίασης του δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκροτεί ένα διπλωματικό σώμα για να επικουρήσει την ΥΠΑ το εκπρόσωπο για την εξωτερική δράση ε, ε, πρέπει να υπάρχει πολιτιστική πολυμορφία, να εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη, να εκπροσωπούνται οι εθνικές εμπειρίες, οι εθνικές παραδόσεις, να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα, αλλά γι' αυτό χρειάζεται ε, συμμετοχή, ισότιμη συμμετοχή όλων. Ε, και θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς λοιπόν θα συγκροτηθεί αυτό το διπλωματικό σώμα. Ε, θα χρησιμοποιηθεί η γραμματεία της Επιτροπής ε, του Συμβουλίου και επιφανείς ε, διπλωμάτες που θα έχουν αποσπαστεί από τα κράτη-μέλη για να στελεχώσουν αυτό το σώμα. Ε, ανεξαρτήτως προέλευσης και μέσω της διοικητικής οδού θα πρέπει να κατοχυρωθεί αναλογική εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών για να λειτουργήσει εύρυθμα αυτό το διπλωματικό σώμα. Ευχαριστώ, Τεζέιρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα στα πλαίσια του ΠΟΕΜ ε, υπέγραψε μια συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής ε, που έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι δασμοί για τις σε μπανανών από αυτές τις χώρες. Ε, και εφιστώ την προσοχή σας στο ότι υπάρχουν εξαιρετικά αρνητικέ επιπτώσεις στους παραγωγούς στη Μαντέιρα και επίσης στις Κανάρες νήσους στην Ισπανία. Αυτά τα τα προϊόντα αυτών των περιοχών, ούτω ή άλλω, λόγω των γεωγραφικών χαρακτηριστικών αυτών των περιοχών, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερε δυσκολίε ε, και τώρα με τη νέα συμφωνία ε, απειλείται η ίδια η ανάπτυξη των περιοχών. Θα πρέπει να ε, προστατεύσουμε τη θέση των παραγωγών, των παραγωγών τη Μαδέιρα, γιατί με αυτήν τη νέα συμφωνία θα πλημμυρίσει η αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση με μπανάνε από τι χώρε τη Λατινική Αμερική και όχι από τι τις υπερπεριφερειακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Childers. Πριν από ένα χρόνο η SR Technics εταιρεία συντήρησης αεροσκαφών έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου για να αντισταθμιστούν αυτές οι απώλειες και σε δουλειές το 2009 ζητήσαμε ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο καταπολέμησης της παγκοσμιοποίησης. Όμως το απέρριψε η Κομισιόν ως μη πλήρες το αίτημα και δεν έχει μπορέσει πέντε μήνες να συμπληρώσει μία αίτηση η κυβέρνηση της Ιρλανδίας. Δεν ξέρω, είχε δουλειές. Μπορεί να την απασχολούσε βεβαίως η οικονομική καταστροφή την οποία προκάλεσε η ίδια και δεν μπορεί να συμπληρώσει ένα έντυπο αίτησης το οποίο θα σώσει και θα αλλάξει εκατοντάδες ζωές και παραμένει σε ένα σιρτάρι. Αν ήταν κάποιος κοινικός μπορεί βεβαίως να σκεφτεί πως το κάνει αυτό η κυβέρνηση γιατί θα πρέπει να συγχρηματοδοτήσει και αυτή. Σας ευχαριστώ. Τελείωσε ο χρόνος σας. Ο κύριος Κουμουτσάκος κατόπιν. Δεν είναι εδώ από ό,τι φαίνεται, οπότε ο κύριο Σαζάδα. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, απευθύνομαι σε εσά κυρίως όμως τον κύριο Ποτότσνικ για ένα θέμα περιβαλλοντικό και μάλιστα μιλάω για την οδηγία 202 49 που αφορά τον περιβαλλοντική επιβάρυνση, τον θόρυβο δηλαδή από αυτοκινητόδρομους και θα πρέπει βεβαίως να υπάρξουν αυτά τα φράγματα του θορύβου που βεβαίως καταστρέφουν κάπως το τοπίο αλλά οδηγούν και αυτά σε έναν επιπλέον κίνδυνο Οπότε μιλάμε για ένα πρόβλημα υγείας βεβαίως και ε, κίνδυνο για την ζωή. Οπότε θέλω να παρακαλέσω τον κύριο και να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία εδώ πέρα. Για να τηρηθεί η οδηγία. Στόκες. Κύριε Πρόεδρε, στη γη του Μιλόσεβιτς, στην Βοηβοδίνα, ξυλοκοπούνται οι Ούγγροι που υπάρχουν εκεί πέρα και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. 400.000 Ούγγροι ζούσαν στη Βοηβοδίνα, ένα τρίτο του πληθυσμού, αλλά τους εξανάγκασαν να φύγουν και εγκαταστάθηκαν εκεί έπικοι. Οπότε μειώθηκε ο αριθμός τους και έφτασε τις 290.000. Η ξυλοδαρμή, λοιπόν των μειονοτήτων έγιναν από τις διαβόητες μυστικές υπηρεσίες των Σέρβων που έδιραν και τους Αλβανούς όπως πολύ καλά ξέρετε. Πρέπει λοιπόν γρήγορα να σταματήσουμε αυτή την τρομοκρατία και εάν είναι να μιλάμε δηλαδή για ένταξη της Σερβίας πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων θα είναι και η αποζημίωση των δεκάδων χιλιάδων θυμάτων αυτής της ε, γενοκτονίας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σενιζίν. Παρακαλώ, κυρία Σενιζίν. Pani Przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Kobiety są niedostatecznie οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στον τομέα της έρευνας. Ε, στην Ευρώπη 30% είναι των επιστημόνων που είναι γυναίκες. Και ε, ε, στην Πολωνία μόνο 7% των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων είναι γυναίκες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να κινηθούμε για να προαγαγούμε το ρόλο των γυναικών στον τομέα της έρευνας. Γίνεται μια σχετική μελέτη από ένα πολωνικό Ινστιτούτο για να κάνουμε κάτι κατά της ε, ε, διάκρισης, διακριτικής αυτής μεταχείρισης Χρειάζεται βέβαια βοήθεια ε, ο οργανισμός που δρομολόγησε αυτή τη μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό απευθύνω έκκληση γι' αυτό προς την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Higgins κατόπιν. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως έλεγα λοιπόν, χάρηκα που άκουσα πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει την οδηγία κάτι το οποίο με ικανοποιεί γιατί εδώ πέρα εστιάζουμε πραγματικά στις αδυναμίες δεν υπάρχει κάποια προστασία στην οδηγία αυτή για ανθρώπους οι οποίοι αγοράζουν ε, γη ή ταξιδεύουν εκτός Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Η μεγάλη αδυναμία αυτής της οδηγίας ε, χαίρομαι ε, που μπορώ να πω πως ε, ο πρώην Επίτροπος ε, χάρηκε για την νέα αυτή οδηγία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριος Πάσκου, τώρα τελευταίος ομιλητής. Πριν από 20 χρόνια πέθαναν οι Ρουμάνοι για την ελευθερία και για την παιδεία. Υπήρχε στενότατος πολιτικός έλεγχος και μετά τις θυσίες τους ε, ε, απέκτησαν την ελευθερία τους ε, τα πανεπιστήμια και έκτοτε τη χαίρονται. Οπότε θα ήταν ηρωνικό αν η τωρινή απόπειρα του Υπουργείου Παιδείας της Ρουμανίας να εγκρίνει την νομοθεσία για να επαναπολίσει πολιτικοποιήσει το σύστημα τελικά πετύχει. Ε, θα πρέπει να ο, ο ίδιος ο Υπουργός ε, να τοποθετηθεί να μην, για να μην χρησιμοποιηθούν αυθαίρετα κριτήρια. Ε, εγώ είμαι καθηγητής και βουλευτή ε, και απευθύνομαι στου ε, συναδέλφου μου τόσο ώστε να εκθέσουν αυτή την παράνομη πρακτική που σαφέστατα αντιτίθεται στην στρατηγική τη Λισαβόνα ε, για την παιδεία. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε να γίνεται κάτι τέτοιο σε κράτο μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Σα ευχαριστώ. Πραγματικά τελειώσαμε με αυτό το σημείο τη Μέση Διάταξη. Σας ευχαριστώ για την κατανοησή σα, για την πειθαρχία που έπρεπε να επιδείξουμε και ελπίζω όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα